κατέθεσε αιτήματα για τις ε, υποψηφιότητες και τις αλλαγές, τις ε, τροποποίησεις που θέλει να γίνουν σε επιτροπές και αντιπροσωπείες θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά και αν δεν σημειωθούν ενστάσεις κατά των ε, αιτήματων αυτών θα θεωρηθούν εγκεκριμένες οι αλλαγές αυτές. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να περάσω στο επόμενο σημείο της ημερήσιας